Pan Przewodniczący! Koleżanki i koledzy, Panie i Panowie. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Mam że